και τα σχέδια αυτά δεν ευόδωσαν. Στη Ρωσία έχουν και λένε ότι η μικρή Φιλανδία ξεκίνησε το πόλεμο αυτό, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη προκαθοριστεί οι σφαίρες επιρροής. Από αυτά λοιπόν θα πρέπει να ενταχτούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρο. Λοτόφσκι. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η, ε, το επίσημο ρωσικό αφήγημα για, ε, για τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν στόχο όχι μόνο να αποστρέψουν την προσοχή από τις ευθύνε του Σοβιετικού Συνδέσμου για την πρόκληση αυτής της διαμάχης, αλλά κυρίως θέλουν να σπείρουν ζυζάνια στην παγκόσμια κοινότητα. Και ιδιαίτερα ενισχυτικέ είναι οι μορφέ τη Ρωσία προ την Πολωνία, που ήταν η χώρα με τα περισσότερα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μάλιστα δεν θα είχαμε δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο στις 23 δεν υπογραφόταν το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο της Μη Επίθεσης. Φαίνεται ότι δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη αυτό το γεγονός ε, ο Πούτιν. Και αν μια χώρα δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες των εγκλημάτων της, αλλά προσπαθεί να επιρρύψει άλλου ευθύνες, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος εταίρος στο διεθνές προσκήνιο. Ε, το ψέμα ξεκίνησε και στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία αυτά τα ψέματα δείχνουν την ποιότητα της Ρωσίας. Αλλά ε, δεν ε, ρίχνουν φως στο ποιος ήταν πραγματικός υπεύθυνο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σλωτόφσκι. Ε, κύριε Αλεξάνδρου να έχετε το λόγο. οφείλουμε να καταδικάσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια του Πούτινγκ ε, να ε, δώσει άφεση αμαρτιών στην Ρωσία για ό,τι έγινε ε, στη διάρκεια του πολέμου και μετά. Η τραγωδία της Βουλγαρίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1944 όταν ε, κήρυξε πόλεμο στην Βουλγαρία η Σοβιετική Ένωση και μετά την απελευθέρωση συνεχίστηκε το εγκληματικό κομμουνιστικό καθεστώς και η ελίτ ε, του κράτους ε, άνοιξε στρατόπεδα ε, συγκέντρωσης, παράνομα δικαστήρια κλπ. Επομένως η Ρωσία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από την Πολωνία, από τα χώρες της Βαλτικής αλλά και από τη Βουλγαρία. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε οποιαδήποτε επιρροή του Κρεμλίνου ε, θα πρέπει να κρατήσουμε σταθερή σχέση και ευελπιστώ ότι ε, φέτος ε, διακόπτεται το μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Γιουρντάνοφ. Ο κύριος Βιτάνοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τον προηγούμενο Σεπτέμβρη Τούτο το Κοινοβούλιο ενέκρινε ε, ψήφισμα για το μέλλον της Ευρώπης και την ιστορία της. Ε, έγινε αναφορά όμως ε, ναι στο σύμφωνο Ρίβεντρον Μολότοφ αλλά όχι στον φασισμό και τον ρόλο του καθώς και στον ρόλο του κομμουνισμού. Εμείς δεν είναι δυνατόν να ε, το να πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε καμία ε, σχέση ανάμεσα στον Χίτλερ ε, και την Ρωσία. Και εξάλλου εδώ δεν μιλάμε για την Ρωσία, μιλάμε για τη δικιά μας ιστορία, δεν μιλάμε για προπαγάνδα, μιλάμε για αυτά που ζήσαμε εμείς. Ε, θέλουμε ε, να ρίξουμε άπλετο φως σε όλα τα εγκλήματα τα οποία έγιναν ε, κατά της ε, ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βιτάνοφ. Επόμενος ομιλητής, έχουμε σπάτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν πραγματικά φρικτά γεγονότα και η γενοκτονία, ε, το ολοκαύτωμα ή ε, το γεγονός ότι πολλές χώρες της Ευρώπης έχασαν την ανεξαρτησία τους. Αυτό προκάλεσε μεγάλη οδύνη και πολλές είναι οι χώρες οι οποίες καταπιέστηκαν είτε από την ναζιστική Γερμανία είτε από τον κομμουνισμό ο Στάλιν και ο Χίτλερ ήταν δικτάτορες και δεν είναι δυνατόν να προσπαθούν ορισμένοι να βρουν ελαφρυντικά ε, στον Στάλιν και τον Χίτλερ ε, γιατί εξαιτίας τους ε, χιλιάδες επί χιλιάδων άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ε, σιγά σιγά ε, ε, χάνονται και αυτοί που είχαν ζήσει και είχαν προσωπικές εμπειρίες από όλα αυτά τα γεγονότα. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει η νέα γενιά, τι συνέβη πραγματικά και τι, πώς οδηγήθηκαν αυτά τα καθεστώτα υπό τον Στάλιν και τον Χίτλερ σε αυτές τις φρικαλαιότητες. θα, δεν είναι δυνατόν να ξεχνούμε την ιστορία και να δικαιολογούμε εγκλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πάιτ. Μάρκο Τρεώστο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ο χειρότερος ε, τρόπος, η χειρότερη μορφή ιστορικής τρέβλωσης ε, ε, είναι η λύθη. Είναι πολλοί αυτοί που ξέχασαν ή υποχρώνονται να ξεχάσουν τα όσα πέρασαν οι Ιταλοί, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εδάφη στην Ίστρια και στο Φιούμε. Ε, δεν είναι δυνατόν όμως να ξεχνάμε κομμουνιστές του τρίτου, ε, χιλι, της τρίτης χιλιετίας ε, εξακολουθούν να ονομάζουν ε, φασιστικό το καθεστώς ε, της ε, Ιταλίας που όμως υπέφερε τα πάνδυνα στη διάρκεια αυτών των γεγονότων. Γίνεται και μια προσπάθεια φιλοσοφικής εξήγησης ο Τζανπάολο Πάνσα έχει γράψει ένα βιβλίο ε, το οποίο λέγεται «Εχμάλωτη τη σιωπή» ε, και που ε, αναφέρεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο η Ιταλική αριστερά αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα. Και ο Σέντζο Ματαρέλα εχμάλωτος τη σιωπή» ήταν γιατί πραγματικά δέχτηκε την διαστρέβλωση της ιστορίας και δέχτηκε την λύθη αυτών των σημαντικών γεγονότων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δρεώστο. Ο κύριος Ραφαέλ Στανκανέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε δράττουμε τη ευκαιρία ε, αυτής της πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση για την στρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας ε, για να αναφερθώ στον Ζαν Πάολο Πάντσα, ε, έγκριτο δημοσιογράφο ο Ιταλό που δεν είχε, ήταν, ανήκε στην αριστερά αλλά χωρίς να ανήκει σε συγκεκριμένο κόμμα διαβάζοντας ξανά ε, κάποιες από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορίες, ε, ε, σελίδες της ιστορίας της Ιταλίας τον προηγούμενο αιώνα, έγραψε ένα άρθρο όπου αναφερόταν στα εγκλήματα των παρτιζάνων, των κομμουνιστών ανταρτών μετά το 1945 που καλύφθηκαν από την αριστερά και από ορισμένε πολιτικές ομάδες και δυνάμεις οι οποίες αρέσκονται στο να αυτοαποκαλούν είναι προοδευτικές και δημοκρατικές. Ε, ε, πρόκειται για ε, συμβάντα, για γεγονότα τα οποία έγιναν είτε στη διάρκεια είτε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι δυνατόν όμως να χρησιμοποιούμε την ιστορία για λόγους ιστορικούς. Δεν είναι δυνατόν αυτό να το επιτρέψουμε ξανά να συμβεί. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τόμακ. Ευχαριστώ. Πέρυσι καταρτήσαμε ένα ψήφισμα στο οποίο καταδικάσαμε το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο μία επίθεση μεταξύ δύο τυράννων που οδήγησε στην κατοχή των χωρών της Βαλτικής, στην εισβολή στην Πολωνία και στη χώρα μου την Ρουμανία. Ε, η πατρίδα μου έχασε λόγω του συμφώνου αυτού εδάφη που δεν τα ανέκτησε ποτέ. Επίσης, ε, εγώ γεννήθηκα σε μια περιοχή που προσαρτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και ακόμη ε, οι Ρουμάνοι της Βεσσαραβίας υφίστανται την προπαγάνδα του καθεστώτος του Πούτιν. Θα πρέπει να πούμε στους πολιτικούς ηθήνοντες της Μόσχας να σταματήσουν την προπαγάνδα τους Επίσης υπάρχει απαγόρευση εισόδου μα ε, στη Ρωσία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την αλήθεια για να διαφυλάξουμε τη μνήμη των προγόνων μας. Σας ευχαριστώ κύριε Τόμακ. Το λόγο έχει ο κύριο ε, Ρουί Ντεβέσα. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση είναι επίκαιρη γιατί έγινε μια απόπειρα πλαστογράφηση τη ιστορία και στρέβλωση τη ιστορία, κάτι που συμβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά. Σήμερα το πρωί, στο, στην Ολομέλη, η κυρία Βίτεκομπ του κόμματο του Brexit είπε ότι το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και ότι αν δεν είχαμε προχωρήσει στην ένταξη θα ήταν ακόμη μαζί μα η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι λάθο. Ε, ε, από την αρχή ήταν ε, υπερεθνικό σχέδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ο ίδιος ο Σούμαν είπε ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα για, μια, για ένα φεντεραλισμό, για μια ομοσπονδία στην Ευρώπη. Ήδη από το 1959, οπότε ήταν τελείως ψέμα αυτά που μας είπε η κυρία Βίτεκομπ. Θα πρέπει λοιπόν όταν βλέπουμε την ιστορία να μην βλέπουμε μόνο τις φρικαλαιότητες που διαπραξαν οι άλλοι και να θελοτυφλούμε στη, στα λάθη των προγόνων μας. Θα πρέπει να δούμε και τα καλά και τις τραγωδίες. Αυτά είναι τμήματα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Σας ευχαριστώ κύριε Ρουσδεβέσα. Το λόγο έχει ο κύριος Πέτρος Αουστρεβίτσιους. Ιστορία τάμπα πολίτικος Πρόεδρε, συνάδελφοι, στα χέρια των εθνικιστών η ιστορία γίνεται πολιτικό εργαλείο και ξαναγράφεται στη Ρωσία. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να στρέψουν τους Ρώσους κατά των ευρωπαϊκών κρατών και για να τους αποσπάσουν την προσοχή από τα τρέχοντα προβλήματά τους. Και αυτά προφανώς ε, απαρνούνται την αλήθεια στην... Λαμβάνεται απόφαση στην παρούσα φάση από το δικαστήριο για την ε, υπόθεση Δημήτροφα. Σε ό,τι αφορά την ε, μνήμη των ε, θυμάτων, των εκατομμυρίων θυμάτων που πολέμησαν κατά του Στάλιν. Τα σταλινιστικά λοιπόν αυτά τα θύματα Ακούσαμε από επίσημες πηγές ότι δεν επρόκειτο για τάφους ε, των θυμάτων του σταλινισμού, αλλά τάφους τάχα των ε, δολοφονηθέντων από το φιλανδικό στρατό. Ο Πούτιν λοιπόν ε, χρησιμοποιεί τέτοιε σταλινιστικές μεθόδους και για να σβήσει τη μνήμη των θυμάτων. Και από την παραποίηση αυτή της ιστορίας καθίσταται σαφές ότι προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε την ιστορία του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Στρεβίτσιος. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Μπίγνιχ Κούσμιουκ. Ευχαριστώ. Κυρία Επιτροπέ, ε, το Σεπτέμβριο του 2019, στην 20η επέτειο της, του ξεσπάσματο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υιοθετήσαμε ψήφισμα ε, δηλώνοντας απερίφραστα ότι το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο Μη Επίθεση της 23 η 8 του 1939, το γνωστό σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, με το συμπληρωματικό ε, πρωτόκολλο, οδήγησε στο διαμελισμό ε, της χώρας και την, το διαμοιρασμό των ζωνών επιρροής και ε, άμεσα οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα το 1 Σεπτεμβρίου ε, ε, η Πολωνία δέχτηκε πρώτα την επίθεση της Γερμανίας και λίγες μέρες μετά την επίθεση του Σοβιετικού στρατού. Ακολούθησαν επιθέσεις σε γειτονικέ χώρες. Και μάλιστα δημοσίω ο Πούτιν αμφισβήτησε αυτά τα ιστορικά γεγονότα επανειλημμένω, προσπαθώντα να επιρρύψει στην Πολωνία ευθύνε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο ακόμη μια φορά να στυλιτεύσει την απόπειρα πλαστογράφηση και στρέβλωση τη ιστορία, αποκρύβοντα τα σοβιετικά, στα ελληνιστικά εγκλήματα και την ευθύνη του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτή την απόπειρα ε, του Πούτιν για τη στρέβλωση της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Κούσμικ. Ο Πέτερ Πόλακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Στις 21 Ιανουαρίου έχουμε την 75η επέτειο της απελευθέρωσης του Auschwitz, ναζιστικό στρατόπεδο όπου έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια αθώοι. Άνθρωποι εντελώς ε, αθώοι και άμαχοι. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε εκ νέου είναι ότι δεν υπάρχουν ε, ούτε ανώτεροι ούτε κατώτεροι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν ανώτερε ράτσες. Και εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή του επειδή ήταν Εβραίοι, επειδή ήταν Ρωμά. Αν είχαν κερδίσει τον πόλεμο οι Νάζοι, δεν θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα, γιατί είμαι Ρωμά και είναι ντροπή το γεγονό ότι Εξακολουθούν να υπάρχουν φασίστες ε, εδώ στο Κοινοβούλιο που αρνούνται το ολοκαύτωμα. Το ολοκαύτωμα έλαβε χώρα και αυτά τα τραγικά περιστατικά δεν μπορείτε να τα παραποιείτε. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχασαν ε, το, τη ζωή τους ε, άνθρωποι επειδή δεν μίλησαν, επειδή ήμουν και σιώπησαν. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να φωνάξουμε κατά των φασιστών. Δεν μπορούμε να σιωπούμε. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το μίσος, γιατί το μίσος είναι ο δρόμος προς την κόλαση. Ευχαριστούμε κύριε Πολάκ. Το λόγο έχει Ρούζα Τόμασιτς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος άφησε ανεξίτηλα ίχνη στην Ευρώπη. Σήμερα, παρόλο που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, ζούμε εν ειρήνη ε, και σε αλληλοσεβασμό, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι συνέβη και ποια ήταν η θέση μας πριν και μετά τον πόλεμο. Δεν ήταν ισότιμη η θέση μας. Μερικοί είχαν υπεριαλιστικές φιλοδοξίες. Άλλοι επιδίωξαν λύση εθνικών ζητημάτων. Άλλοι αμήνθηκαν, υπερασπίστηκαν τις πατρίδες τους. Και άλλοι απλώς ήταν αντάλλαγμα. Ε, μερικοί ε, όντως απελευθερώθηκαν από τον τρόμο, από τις δυτικές ε, ε, δυνάμεις και άλλοι έμειναν εχμάλωτοι των κομμουνιστών. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος καλύπτει μια σειρά τοπικών σειράξεων που είχαν ένα κοινό υπόβαθρο. Αν τα λάβουμε όλα αυτά, είναι σαφές γιατί είναι σημαντική η μνήμη για τα γεγονότα αυτά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει να καταδικάζουμε τους εγκληματίες και την εγκληματική ιδεολογία και οποιοδήποτε ολοκληρωτισμός, είτε είναι ναζιστικός, είτε φασιστικός, είτε κομμουνιστικός, θα πρέπει να καταδικαστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Τόμασιτς. Η κυρία Γιοκνεβιτσιανέ. Σε ό,τι αφορά τον Ρώσο πρόεδρο, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το γεγονός ότι έχει κάνει μεγάλη διαφήμιση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πούτιν λοιπόν βασίζεται σε ε, αρχείο και υλικό το οποίο εδώ και καιρό δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Θα ήθελα να σας στήσω τον κύριο Πούτιν να δημοσιεύσει όλο το αρχείο από την εποχή του Στάλιν. Όλο το υλικό αυτό. Και μάλιστα να το διαθέσει στην ε, κοινή γνώμη. Γιατί η κοινή γνώμη έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι συνέβησε στους Εβραίους και ο Πούτιν θα πρέπει να επιστρέψει στη Λιθουανία τα κλεμμένα αρχεία που, του 1991. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο κόκκινος στρατός είχε δικαίωμα ανοιχτά να βιάζει γυναίκες και να καταστρέφει αμάχους, να εκτελεί αμάχους. Θα πρέπει να ξέρει η κοινή γνώμη ότι άνοιγαν σκυλιά των αγίων Antaisin sitten seuraavaksi puheenvuoron η Ντούρις Νίκολσονόβα, για ένα λεπτό. τον 20ο αιώνα τα ναζιστικά καθεστώτα εκτέλεσαν εκατομμύρια ανθρώπους και αυτό αποτελεί μια προειδοποίηση για τις επόμενες γενναίες. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Στην χώρα μου προωθούνται οι νεοφασιστές και έχουν μπει στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ένας πολιτικός ο οποίος ε, υποστηρίζει κομμουνιστικές ιδεολογίες είναι επικεφαλής του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά ντροπή. Εγώ ντρέπομαι και θα πρέπει να εξετάσουμε τα βαθύτερα αίτια για την υποστήριξη των ακροδεξιών. Η διαφθορά, η έλλειψη εκπαίδευσης και παιδείας και πολιτισμού και αυτά οδηγούν τους πολιτικούς να αμφισβητούν το ολοκαύτωμα και να σπέρνουν το μίσος. Και αυτό οδηγεί στην επιδημία του εξτρεμισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Σόνοβα. Τώρα κυρία Σόντροβα. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι το σύμφωνο Ρίβεντροφ Μολότοφ αποτελεί μια υπενθύμηση για το τι συνέβησε Και αυτό δίνει δικαίωμα να θεωρήσουμε και του Ρώσου εισβολεί, παρά το γεγονό ότι συνέβαλαν στην πτώση τη γερμανικού καθεστώτο, του ναζιστικού καθεστώτο. Και έτσι λοιπόν μα κατηγορούν ότι είμαστε. Κατηγορούν την Πολωνία ότι ήταν ε, χώρα που επιτέθηκε. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό σφάλμα. Δεν είμαστε οι ε, ρατσιστές. Ε, θέλουμε να εκφράσουμε το γεγονός ότι είμαστε ενάντια στα ιστορικά ψέματα του Προέδρου Πούτιν. Δεν θέλουμε ε, να ξαναέρθει δικτατορία ή πόλεμος στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να το υπενθυμίζουμε διαρκώς ε, για να το ακούν και οι μελλοντικέ γενναίες. Σας ευχαριστώ κυρία Σόιντροβα. Ο τελευταίος ε, ομιλητής στη συζήτηση αυτή είναι ο κύριος Αρσαλέχος. Για ένα λεπτό. Όταν μιλούμε για το παρελθόν σε ένα θεσμικό όργανο σαν το δικό μας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν είμαστε ιστορικοί. Είμαστε όμως προϊόν της ιστορίας. Και για να μείνουμε πιστοί σε αυτή την ιστορία, δεν μπορούμε να ξεχνούμε, θυμίζοντας το στίχο του Χόρχε Λουίς του Αργεντίνου ποιητή, ότι την Ευρώπη δεν την ένωσε η αγάπη, αλλά η φρίκη. Η φρίκη του ολοκαυτώματος, του ολέθρου, η φρίκη του ρατσιστικού εθνικισμού που έχει ακόμη απογόνους αυτό το κοινοβούλιο και ε, έχουν το θράσος να δίνουν μαθήματα σε μια μεγάλη δημοκρατία όπως η Ισπανία. Η, φρά, φρίκη του ναζισμού, του κομμουνισμού, η φρίκη του Μολότοφ και του Φορίμπετροπ. Γι' αυτό και θα πρέπει να επαγρυπνούμε απέναντι στις απόπειρες στρέβλωσης της ευρωπαϊκής ιστορίας, στις απόπειρες να αθωθούν τα μαζικά εγκλήματα των στρατοπέδων εξόντωση στο Ναζί ή του Σοβιετικού Γκουλάκ. Γιατί η οδύνη των Ευρωπαίων στα χέρια αυτών των εγκληματικών καθεστώτων δεν είναι υποδιαπραγμάτευση είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατασκευάστηκε ως σχέδιο ειρήνης και ελευθερίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Θαρθαλέχος. Και τώρα για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση θα δώσω το λόγο ε, στην Επιτροπή, στην κυρία Γιούροβα και μετά στο Συμβούλιο. Η κυρία Γιούροβα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Βουλευτέ. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω εν συμπεράσματι ότι εάν ε, μια χώρα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί ή προσπαθήσει να διαστρεβλώσει μέσω εσφαλμένων πληροφοριών την ιστορία, η Κομισιόν θα λάβει αμέσως ε, μέτρα. Ε, το ίδιο θα κάνει και για να διατηρηθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Ούτως ή άλλως ε, το ιδεώδες ε, του αυταρχισμού ε, δεν αφορά μονάχα τον ναζισμό ή τον κομμουνισμό, αλλά ανθρώπους για τους οποίους ο διαχωρισμός μεταξύ του πραγματικού και της μυθοπλασίας και ο διαχωρισμός ανάμεσα του πραγματικού και του μη πραγματικού δεν υφίσταται πλέον. Εγώ θέλω βάσει της εντολής μου και της αποστολής μου να ενισχύσω την την ανθεκτικότητα των μέσων, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, ε, τα οποία θα πρέπει να παραμένουν προσκολλημένα πάντοτε στα πραγματικά περιστατικά, τα πραγματικά γεγονότα και την αλήθεια. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να μπορεί να γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα στο αληθές και το ψευδές μην λησμονούμε ότι ε, πρόσφατα γιορτάσαμε την 70η επέτειο από το τέλος ε, του πιο αιματηρού πολέμου στην ιστορία της Ευρώπης. Ε, δεν θέλουμε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και ούτε θέλουμε τα θύματα να, φορέσουν το, να τους φορέσουμε το προσωπείο των κατέχοντων. Κυρίε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει πολλά να διδαχθούμε από την ιστορία μας, τους καιρούς αυτούς που οι κοινέ μας αρχές είναι έθραυστες και θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να στηριζόμαστε σε κοινέ αξίες και αμοιβαία κατανόηση για τη θέση μας και συνειδητοποίηση της ιστορίας της Ευρώπης, ακόμη και του ολοκληρωτισμού που είναι έτοιμα αυτής της ιστορίας. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δηλώση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις ενεξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Ουγγαρία. Εξ ονόματος του Συμβουλίου το λόγο έχει η κυρία Μπρίνιεκ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι πυλώνας των κοινών μας αξιών και βρίσκεται στην καρδιά της Ένωσης μας και πειράζει άμεσα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και το περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις μας δραστηριοποιούνται. Κάποιες αδυναμίες στον τομέα αυτό καθιστούν την κοινωνία μας και την Ένωσή μας πολύ πιο έθραυστη και εσωτερικά και εξωτερικά. Ο ίδιος ο ιστός των κοινωνιών μας ε, ε, στηρίζεται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά τα στοιχεία είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και ε, αμοιβαία ενεργοποιούνται και ενισχύονται. Και τίποτα δεν είναι χωρίς τα άλλα. Το άρθρο 2.1 για το άρθρο 7.1 συνεχίζονται οι διαδικασίες για την Ουγγαρία και την Πολωνία. Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά για την Ουγγαρία που ενεργοποιήθηκε μετά την πρόσφατη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου 2018, έγιναν δύο ακροάσει το προηγούμενο εξάμεινο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στι 16 Σεπτεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου του 2019. Η πρώτη ακρόαση ήταν γενικού χαρακτήρα και κάλυψε όλα τα θέματα που περιλάμβανε η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δεύτερη ακρόαση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα θέματα. Ελευθερία έκφραση, πολυφωνία των μέσων μαζική ενημέρωση, ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακή ελευθερία και ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία. Όπω αναφέρεται στη διαδικασία για τι ακροάσει του άρθρου 7, και κρίθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο, η Φιλανδική Προεδρία ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαδικασία αυτή και μετέφερε ε, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ακρόαση για την Ουγγαρία. Στι 4 ε, Σεπτεμβρίου πριν την ακρόαση, μαζί με τη Κροατική και τη γερμανική ε, προεδρία, του τρίτου των Προεδριών, συναντήσαμε τον πρόεδρο τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, που είναι και εισηγητή για το θέμα αυτό. Στι 10, 10 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τη δεύτερη ακρόαση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών. Ε, μια άτυπη συνάντηση Υπουργών και Κοινοβουλίου έλαβε χώρα. Και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε την αιτιολογημένη του πρόταση και τι απόψει του για τι πρόσφατε εξελίξει στην Ουγγαρία. Κατά τη διάρκεια τη κρατική Προεδρία, είναι πρόθεσή μα να συνεχίσουμε να κρατούμε τακτικά ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σε δυνάμει του άρθρου 7 και την διαδικασία που αφορά την Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής, το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμπεριλάβατε το θέμα σχετικά με την Ουγγαρία στη σημερινή ε, ημερήσια διάταξη είναι σημαντικό ε, το κάθε θεσμικό όργανο να τηρεί τον ρόλο του. Στις 8 Νοεμβρίου η πρόεδρος Ουσούλα Βαφόντερ Λάιεν υπενθύμησε ε, εδώ σε τούτη την αίθουσα ότι το κράτος δικαίου αποτελεί το θεμέλιό μας και δεν είναι δυνατόν να υποστεί οποιαδήποτε αλλίωση. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή αυτή παντού και όλες οι χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ε, υπενθύμησε δε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διάλογος και πρόληψη, αλλά ε, και να λαμβάνονται αναπερίπτωση τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την Ουγγαρία. Η Κομισιόν επανειλημμένα ε, έχει ε, αναφερθεί σε σημαντικό προβληματισμό που έχει προκληθεί και βάσει του οποίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 7 παραγράφου 1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 Οπωσδήποτε ε, θα πρέπει όμως οποιαδήποτε δράση να ε, αφορά συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Πιο πρόσφατα η Κομισιόν στη διάρκεια της ακρόασης ε, για την Ουγγαρία στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του μηνός Δεκεμβρίου υπενθύμησε τις αρχές αυτές και εγώ η ίδια αναφέρθηκα σε προβληματισμούς που αφορούν αφορούν την Ουγγαρία και που αναφέρονται διεξοδικά σε πρόσφατη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Ε, το κράτος ε, δικαίου, ε, σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος εγκρίθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο χωρίς όμως πρώτερη διαβούλευση. Αξιολογούμε αυτήν την ομοθεσία που πέρασε την 10η Σεπτεμβρίου του 19. Το Ανώτο Δικαστήριο ε, έβγαλε απόφαση ε, η οποία αφορά ε, την, το αφορά προδικαστικό ερώτημα που είχε υποβληθεί ε, και ε, αφορά ακριβώς τον μηχανισμό του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου. Αυτός ο μηχανισμός αντιμετωπίζει προβλήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν αντίκτυπο γενικότερα στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Επίσης, το προηγούμενο Δεκέμβριο, έξι διεθνείς οργανώσεις δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι από το 2010 η Ουγγρική κυβέρνηση συστηματικά ε, έχει ακυρώσει την πολυφωνία των μέσων ε, ενημέρωσης από τη στιγμή που ε, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται πλέον στα χέρια της κυβέρνησης. Επίσης, το γεγονός ότι πάνω από 400 ε, μέσα ε, διαφορετικού είδους βρίσκονται πλέον ε, στον ίδιο όμιλο holding προφανώς μας δημιουργεί προβλήματα. Είναι θέμα, στοιχείο το οποίο αναφέρεται σε αυτήν την έκθεση. Και βεβαίως μας απασχολεί σε αυτή η κατάσταση όσον αφορά την γενική κατάσταση πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης η ε, προσπάθεια ε, να ε, υπεκφύγει η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού και η αρχή των, που διέπει το μέσα ενημέρωσης να υπεκφύγει όσον αφορά την συζήτηση για τα θέματα αυτά προφανώς δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Επίσης ε, έχει υπάρξει και ένας νέος νόμος ε, ο οποίος ε, έχει υποστεί πολλές επικρίσεις αφορά την επιστημονική έρευνα και τον έχουν επικρίνει πολλές ανεξάρτητες αρχές επιστημονικές και επιστημονικά ακαδημαϊκά συμβούλια. Όσον αφορά τον γενικότερο φάκελο που αφορά αυτές τις εξελίξεις, η Κομισιόν δηλώνει ότι ότι είναι απολύτως διατεθειμένη να λάβει ε, μέτρα όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα και εξελίξεις που έχουν προκύψει ε, στην Ουγγαρία. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει ε, πολλές διαδικασίες επί παραβάση σε σχέση με την Ουγγαρία, οι οποίες σχετίζονται με την ακαδημαϊκή ελευθερία, την, το δικαίωμα σε απόλυτες πληροφορίες, το δικαίωμα της μετακίνησης και άλλο όσον αφορά το εξάμεινο ε, η Κομισιόν ε, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο έχει λάβει συγκεκριμένη ε, γνώση όσον αφορά θέματα διαφοράς, διαφθοράς και προσβασιμότητας του κοινού σε πληροφορίες. Τελειώνω λέγοντας ότι η Κομισιόν παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση, συνεχίζει την αξιολόγηση των στοιχείων που τις έχουν υποβληθεί ε, και θα είναι πάντα στο πλευρό των πολιτών. Των λοιπόν, ομάδων. Ε, για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει η κυρία Μέτσολα για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συζητάμε σήμερα το κράτο δικαίου εκ νέου. Είναι ενσυχητικό το θέμα αυτό ανακύπτει εκ νέου και η τοποθέτηση του ΕΛΚ ήταν πάντα ξεκάθαρη και συνεπείς σε ό,τι αφορά όλες τις χώρες. Δεν θέλουμε το κράτος δικαίου να... Θέλουμε μάλλον να, είναι, να διατηρείται πάντα το κράτος δικαίου με σαφή τρόπο και με διαφανείς διαδικασίες. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό πιστεύαμε και αυτό εξακολουθούμε να πιστεύουμε γιατί χωρίς κράτος δικαίου τα θεσμικά όργανα βλάπτοντα. Δεν υπάρχει υποστήριξη και προστασία του πολίτη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια σημαίνει ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό λοιπόν η Ένωση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουν και να προασπίσουν το κράτος δικαίου. Πάντα θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό των πολιτών, στο πλευρό του δικαίου, στο πλευρό της δικαιοσύνης. Και αυτό δεν θα πρέπει να αμφισβητείται από καμία χώρα, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από κανένα θεσμικό όργανο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να διατηρήσει την αξία και την του κράτους δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου από κάποια χώρα. Οι αξίε στην οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα πρέπει να συνενώνουν τις χώρες και θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα ενισχύουμε τους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την προάσπιση του κράτους δικαίου γιατί οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να έχουμε από τους πολίτες μας. Θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή, θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος θα ισχύει για όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια μέτρα δηλαδή. Όλες οι χώρες θα πρέπει να περνούν από μια τέτοια αξιολόγηση. Έτσι πραγματικά θα εκπροσωπούμε όσους μας εξέλεξαν. Έτσι θα προστατεύσουμε τους πολίτες. Των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει η κυρία Σπούρεκ για δύο λεπτά. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. 17 μήνες έχουν περάσει από την διαδικασία κατά της Ουγγαρίας και από την θέση ισχύ του άρθρου 7. Έχει αλλάξει η κατάσταση στην Ουγγαρία. Τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυριζόταν ότι οι Ουγγρικές αρχές περιόριζαν τις ε, ε, ελευθερίες ε, των μέσων, των πανεπιστημίων και καταπίεζαν τις μειονότητες. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠ εργαζόμαστε για μια έκθεση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία. Και χωρίς όμως την έκθεση είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι ακροάσεις που έγιναν σε ό,τι αφορά το δεν επέφεραν καμία πρόοδο. Αυτό ασφαλώ δεν είναι πρόβλημα μόνο τη Ουγγαρία, γιατί προφανώ αυτό το άρθρο 7 ισχύει και για την κατάσταση στην Πολωνία. Α το παραδεχτούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν έχει δυνατότητα να ανακτήσει και να επαναφέρει το κράτο δικαίου γρήγορα στα κράτη-μέλη. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου για νέου μηχανισμού. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Για την ομάδα Renew Europe το λόγο έχει η κυρία Στρουγκάριου για 1,5 λεπτό. I εδώ θεωρώντας ότι καλωσορίζουμε μεν τις ακροάσεις που διοργάνωσε το Συμβούλιο μας, ανησυχεί η έλλειψη συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλω πραγματικά όμως να συζητήσω τα διαδικαστικά θέματα. αλλά γνώμη. Θέλω να μιλήσω για το γεγονός ότι είναι ντροπή αυτό που κάνετε στη χώρα σας. Την είστε στη χώρα, κύριε Ορμπάν. Είναι ντροπή αυτό που κάνατε για τη θέση που αξίζει να έχει η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην καλλιτεχνική αμα, ελευθερία, στην ε, κοινωνία, κοινότητα των ε, καλλιτεχνών και όλων των πολιτών. Ξέρετε, δεν σα ανάγκασε κανεί να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια επιλογή και μια δέσμευση σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ αξίε. Τι αξίε αυτέ τι οποίε δεν σέβεστε. Δεν σέβεστε την ίδια την επιλογή σα. Ξέρετε ότι η Ουγγαρία αναπτύχθηκε τόσο όμορφα χρησιμοποιώντας ε, τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το ίδιο και η Πολωνία. Και τώρα χτίζεται πραγματικά αυτοκρατορίες μίσους και παραπληροφόρησης και χειραγώγησης χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους. Είσαστε πραγματικά ντροπιαστικός. Και αν δεν υπάρχουν ε, αρκετέ οι διαδικασίε, να τι ε, καθιερώσουμε. Αν δεν υπάρχει η νομοθεσία, να την καταρτήσουμε. Να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε και εσά και οποιονδήποτε άλλο από το να φέρνουν ντροπή στη χώρα τους με τέτοιο τρόπο. Και μια τελευταία σκέψη προς το Συμβούλιο, επιτρέψτε μου. Με τη συνεργασία σας ε, και η διαφάνειά σας ε, δεν βλάπτουν ιδιαίτερα αν είναι προς όφελος των πολιτών και τη Ένωσης των Ευρωπαϊκών Αξιών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των ε, Πρασίνων. Το λόγο έχει η κυρία Ντελμπό Κορφίλ για δύο λεπτά. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της Ουγγαρίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Φιλαδική Προεδρία έκανε επιτέλεσε ένα πολύ σοβαρό, θαραλέο και ε, σημαντικό έργο. Καλή προεργασία για την κρατική προεδρία. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 θα πρέπει να συνεχίσει να ε, ενεργοποιείται κατά της Ουγγαρίας. Ε, κάποια στιγμή η κατάσταση είχε κολλήσει, αλλά χάρη στις ακροάσεις ε, που οργάνωσε η Φιλανδική Προεδρία, διαπιστώσαμε ότι υπήρξε κάποια μικρή πρόοδο. Μια μικρή εξέλιξη, ανεπέστητη, αλλά υπήρξε και ελπίζω και η Κροατική και η Γερμανική Προεδρία να συνεχίσουν το καλό έργο που ξεκίνησαν οι Φιλανδοί. Η ακρόαση ήταν το πρώτο σημαντικό στάδιο της διαδικασίας. Δεν ήταν εύκολο ε, μια χώρα να αξιολογηθεί από άλλες ε, ισότιμες χώρες. Ήταν πολύ εντυπωσιακή διεξαγωγή των ακροάσεων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως και να ε, οργανωθεί και τρίτη ακρόαση για την χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Ίσως θα μπορούσε να είναι το το αντικείμενο τη επόμενη ακρόαση. Κύριε Γιώργο, μιλήσατε για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται κοινοτικά κονδύλια για να διευκολύνεται η συγκέντρωση των ΜΜΕ στην Ουγγαρία. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό. Όπω είπε η κυρία Στρουγκάριου, έχουμε και θεσμικό πρόβλημα εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμη δεν έχει λάβει επίσημα ε, τα απορίσματα των ακροάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση και το ψήφισμα που θα κληθούμε να ε, ψηφίσουμε αύριο αναφέρεται σε δύο διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας και κατά της Πολωνίας. Υπάρχει μια αδικία στη μεταχείριση. Στην περίπτωση της ε, Πολωνίας ε, γίνεται ακρόση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας δεν έχουμε δώσει ακόμη επίσημα τη γνώμη μα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι άτυπε συνεδριάσεις δεν μας αρκούν ούτε μα ικανοποιούν. Δημιουργείται ένα προηγούμενο που δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτή η αδικία θα πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ. Για την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία το λόγο έχει ο κύριος Ριβιέρ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, σε αυτήν την περίπτωση της ενεργοποίησης του άρθρου 7 για την Ουγγαρία, στην ουσία το Κοινοβούλιο γίνεται απλώς γραμματέας ε, της ε, Κομισιόν, γιατί εδώ μιλάμε για μια κυρίαρχη χώρα και επομένως το θέμα δεν είναι νομικό, είναι πολιτικό. Η διαδικασία ενάντια σε μια χώρα που, το, της οποίας η κυβέρνηση είναι δημοκρατικά εκλεγμένη, όπως έγινε στην περίπτωση του ε, Πρόεδρου Ορμπάν και μάλιστα επανειλημμένα, ε, ε, πρέπει να θυμίσω ότι περίπου 50% των ψήφων έλαβε η κυβέρνηση Ορμπάν στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτήν την την κατάσταση όσον αφορά τους μετανάστες και αυτό το πρόσχημα του νόμου Stop Soros δεν είναι αστείο. Θα πρέπει τα κράτη να έχουν την δυνατότητα σε διαφάνεια να προχωρούν. Αλλά ακόμα και αυτήν την μεγάλη διαφάνεια τη βρίσκεται αντιδημοκρατική. Εσείς στην ουσία θέλετε να ξεκινήσετε διαδικασία ε, λες και είμαστε όλοι απάτριδες και λες και όλοι ε, υποκύπτουμε ε, στα μεγάλα κεφάλαια. Δεν θα πετύχετε σε αυτήν την διαδικασία και εκ των προτέρων η προσπάθειά σα έχει αποτύχει και χαίρομαι γι' αυτό. Και το λόγο έχει ο κύριος Προκατσίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια φορά και έναν καιρό ε, υπήρχε μία νόμιμη δημοκρατική κυβέρνηση που βγήκε από, προέκυψε από εκλογές που αποφάσισε να αγαπήσει πείσει τι ρίζε πολιτιστικές και θρησκευτικές που είχε ε, και ε, να προστατεύσει τα σύνορα. Αλλά ε, αυτός ο κόκκινος ακάματος φρουρός των συνθήκων, ο Φραντς Τίμερμανς, ενεργοποίησε το άρθρο 7. Συνέβη η ιστορία αυτή στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, αλλά θα μπορούσε να, χρησιμοποιηθεί, να, να συμβεί παντού με την χρήση του άρθρου 7 ε, στην ουσία θέλει ε, η Κομισιόν να χτυπήσει έναν έτσι ώστε να καταλάβουν οι πολλοί. Νομίζω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση και σας το λέω εκ των προτέρων να, ξεκινήσει, να, να προετοιμαστείτε για μια διαδικασία ε, ε, ε άρθρο 7 και για την Ιταλία. Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, το λόγο έχει η κυρία Μπιόρκ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Είμαι υπερήφανη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε θέση για τα τεκτενόμενα στην Ουγγαρία. Και χαίρομαι που ταχθήκαμε υπέρμαχοι της δημοκρατίας των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ε, δυστυχώς η πολυφωνία του τύπου περιορίζεται, η ακαδημαϊκή ελευθερία φημώνεται και για πρώτη φορά έχουμε μεταφορά πανεπιστημίου. Ε, επίσης, ε, η Ουγγαρία επιτίθεται στους μετανάστες και τους στερεί σημαντικά δικαιώματα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ελευθερία των δικαστηρίων, ενώ η νέα νομοθεσία θα φημώσει και τους δικαστές καταπατώντας τη δικαστική ελευθερία. Η χρήση επίσης των γεωργικών ενισχύσεων τελικά πήγε στις, πήγαν στις τσέπες των ολιγαρχών που ουσιαστικά συνεργάζονται με την εξουσία. Υπάρχει διαπλοκή συμφερόντων. Γίνεται μία απόπειρα να φημωθεί και η αντιπολίτευση, κάτι που είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε σεβασμός θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Πολλοί κόσμοι στην Ουγγαρία διαφωνεί με την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν, υπάρχουν ε, Ούγγροι που είναι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, των μεταναστών, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ του κράτους δικαίου. Και αν ε, κινητοποιηθούν όλοι αυτοί οι Ούγγροι πολίτε ίσω καταφέρουν κάτι, αλλά δεν μπορούμε εμεί να σιωπούμε και να μένουμε σταυρωμένα χέρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση ω έχει. Ευχαριστούμε τη Φιλανδική Προεδρία για την ενεργοποίηση τη διαδικασία του άρθρου 7 κατά τη Ουγγαρία. Στην περίπτωση τη Πολωνία όμω δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Έχει πάρει κακό δρόμο η διαδικασία. Θέλουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να προασπίσουμε το κράτο δικαίου. Ειδικά τώρα που θα συζητήσουμε και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει τώρα να θέσουμε αυστηρές προϋποθέσεις για να βάλουν μυαλό αυτοί που παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Το λόγο έχει η κυρία Φεράρα για 1,5 λεπτό, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μεταξύ των ε, κοινών αρχών επί των οποίων βασίζεται ε, το, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος δικαίου αποτελεί το επιστέσγασμα, την κορονίδα των δικαιωμάτων και των εξουσιών. Μία κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να διευρύνει την εξουσία ε, δυναμητίζοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία έκφρασης δεν είναι δυνατόν να κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι έχει εκλεγεί δημοκρατικά και θύματα δεν είναι μονάχα οι πολίτες ε, οι οποίοι βλέπουν να συρρυκνούνται τα δικαιώματά τους ε, ε, αλλά και οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και η εμπιστοσύνη των πολιτών στις κοινέ αρχές. Και στην περίπτωση της Ουγγαρίας αλλά και αλλού μπορεί να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ωστόσο η διαδικασία της του... του άρθρου 7 παράγραφος 1 ε, δεν δίνουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις ε, και επομένως δεν είναι προσήκον το άρθρο αυτό. Ε, και η κυβέρνηση Ορμπάν είναι τόσο ε, σίγουρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ε, τιμωρία που συνεχίζει την ίδια πορεία. πορεία. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ακέραιος και ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός. Ένας οργανισμός ο οποίος θα παρακολουθεί και την, τις διαδικασίες που αφορούν το κράτος δικαίου και της κυρώσεις και την επιβολή των κυρώσεων. Η, η κυρία Γιάροκα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε που η συζήτηση για την Ουγγαρία έχει γίνει μαϊδανός στην ημερήσια διάταξη Ολομέλειας. Κάθε τρεις και λίγο ε, τη βλέπουμε στο πρόγραμμά μας. Βέβαια, η συζήτηση αυτή δεν αφορά πραγματικά περιστατικά, αλλά ένα πολιτικό κυνήγι ε, μαγισσών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί αμφισβητούμε την ανεξαρτησία του Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Ακούμε κατηγορίε, αλλά φαίνεται ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Αυτοί που μα κατηγορούν δεν ενδιαφέρονται για την ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία στην Ουγγαρία. Ε, στην Ουγγαρία ισχύει μηδενική ανοχή κατά τη ε, διαφθοράς. Έχουμε πολύ καλή στρατηγική από την άποψη αυτή, αλλά φαίνεται ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ φαίνεται ότι ενημερώνονται από τα αριστερίζοντα ΜΜΕ, που υποτίθεται ότι καταπιέζονται από την Ουγγρική κυβέρνηση. Εδώ βρισκόμαστε σε μία ακόμη συζήτηση που αντιβαίνει και στο πνεύμα και στο γράμμα της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία νομική διαμάχη δεν μπορεί να διευθετηθεί με μια επιθετική πολιτική συζήτηση. Αυτό είναι το δίδαγμα του κομμουνισμού. Κυρία Γιάροκα, έχετε μια ερώτηση με μπλε κάρτα από την κυρία Ίντβελτ. Τη δέχεστε? Βεβαίως. Κυρία Ίντβελτ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ συνάδελφε, συνάδελφε, μία διόρθωση καταρχήν. Δεν έχουμε συζήτηση για την Ουγγαρία αλλά για την στάση της Ουγγρικής κυβέρνησης. Δεν ταυτίζονται τα δύο. Σας ερωτώ λοιπόν. Είναι σαφέστατος ο τίτλος της συζήτησης. Αγαπητοί συνάδελφε, έχω μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί συνεχίζετε να επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια. Ότι κάνουμε ισχυρισμούς. Μπορώ να ρωτήσω επιτέλους. Θα μου επιτρέψετε να υποβάλω την ερώτησή μου. Παρακαλώ, σεβαστείτε τους κανόνες του Κοινοβουλίου και μην διακόπτετε την ομιλήτρια. Όλα τα ίδια και τα ίδια λέτε. Ότι μας ενημερώνουν τα αριστερίζοντα ΜΜΕ. Τι θα πει αριστερίζοντα ΜΜΕ. Περιλαμβάνεται στα αριστερίζοντα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, την Επιτροπή της Βενετίας, ε, ε, το, ε, τον ΟΑΣΕ. Ε, δεν είναι ανεξάρτητα θεσμικά όργανα η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι όλοι κυριαρχούνται από την αριστερά. Ποια είναι τα αριστερά έψιλον ε που, που αναφέρατε στην ε, παρέμβασή σας. Μισό λεπτό κύριε Γιάρκο για την απάντηση. Μόνο πέντε ΜΚΟ έχουν δώσει αυτές τις πληροφορίες. Το ξέρω γιατί μαζί κάναμε την έκθεση στην Αργεντίνη. Και αυτό ήταν το τμήμα των Ρωμά και διαπιστώσατε ότι και αυτά ήταν ε, ψέματα. Αυτά τα ΜΜΕ σα δίνουν ανακριβείς πληροφορίες. Ελάτε παρακαλώ στην Ουγγαρία να δείτε την κατάσταση με τα ίδια σας τα μάτια. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπάρλεϊ για 1,5 λεπτό. Ähm, Ευχαριστώ. Χτε μόλις ε, ζητήθηκε κατά δική τη ε, Ουγγαρίας ε, από το δικαστήριο. Και αυτό είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο ενδεχομένω να τον γνωρίζει η κυρία Γιάρακά σε ό,τι αφορά και τι καταγγελίε καταγγελίες στο ΜΚΟ για την ε, παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Α είμαστε λοιπόν ειλικρινεί ότι η διαδικασία του άρθρου 7 κατά τη Πολωνία και κατά τη Ουγγαρία έχει φτάσει σε αντιέξοδο. Όταν ε, καταρτίστηκε αυτή η διαδικασία, δεν είχαν φανταστεί οι προπάτορε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα υπήρχαν δύο κράτη-μέλη τα οποία θα, δεν θα συμμορφούνταν με τι ε, προδιαγραφέ αυτέ. Και αυτό ακριβώ έγινε χθε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Ουγγαρίας, ε, το ΕΛΚ ε, εδώ και χρόνια έχει διστάζει να χρησιμοποιήσει τα ξεκάθαρα λόγια που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει. Έχουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Χρειαζόμαστε πιο πολλά μέτρα. Θα πρέπει να αποτρέψουμε τα καθεστώτα αυτά να αγοράζουν, εξαγοράζουν την υποστήριξη των λαών τους με ευρωπαϊκά χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφείς ε, διατάξεις σε ό,τι αφορά τις ε, οικονομικές ε, συνέπειε που θα πρέπει να έχει η μη συμμόρφωση με τι ευρωπαϊκέ αξίε. Αυτό που είναι σημαντικό ότι δεν προσάπτουμε τίποτα στον κόσμο, στον λαό τη Ουγγαρία, στην κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι φίλοι τη Ευρώπη εκεί και αυτού θα πρέπει να υποστηρίξουμε, να βοηθήσουμε, να δώσουμε μια πλατφόρμα. Το λόγο ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ και πως πολύ από Όπω είπαν πολλοί ευρωβουλευτέ, η, Ουγγρική κυβέρνηση εδώ και μια δεκαετία κλέβει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταρρύπτει το κράτο δικαίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει σοβαρά βήματα για να σταματήσει τη διαδικασία αυτή. Συνεχίζει να δίνει χρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Ουγγρική ελίτ για να α, χτίζει ιδιωτικά ταμεία αντί να χρηματοδοτεί τα σχολεία και άλλε δημόσιε υπηρεσίε η Ουγγρική κυβέρνηση αυτά τα παίρνει στον Και αν παρακολουθεί κανεί τι γίνεται στην Ουγγαρία, διαπιστώνει ότι από τότε που συζητούσαμε τα θέματα αυτά και από την έκθεση σε Αργεντίνη έχουν γίνει και περαιτέρω επιθέσει κατά τη δημοκρατία. Είναι τόσο συνηθισμένοι στο να δρούν ατιμόρυτα που κάνουν και σχόλια κατά των Ούγγρων δεν υπάρχει λοιπόν κανένα όνειδος πλέον. Καταπατούν τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ, αξίες, ενώ εμείς συζητάμε συζήτηση κατά, μετά από συζητήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βασικά σιωπεί σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Και αυτό που πραγματικά λειτουργεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε μπλε κάρτα από τον κύριο Σβέν Σίμον. Τη δέχεστε, κύριε Ντόναντ. Μάλιστα. Κύριε Σβέν, έχετε το λόγο. Για 30 δευτερά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση ότι θα κάνουμε διάκριση, να κάνουμε διάκριση μεταξύ ε, γεγονότων και πολιτικών απόψεων. Γι' αυτό, αγαπητέ κυρία συνάδελφοι, θα ήταν σημαντικό να περιορίσετε στα γεγονότα και στο δίκαιο να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, τεκμηριωμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνείτε μαζί μου. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, για να απαντήσετε. Όπως ε, όλοι είπαν, καταρρύπτονται οι πράξεις από το βάρος όλων των ε, τεκμηρίων, όλων των αποδεκτικών στοιχείων. Δεν μπορούμε να, διακ κάνουμε διάκριση μεταξύ των γεγονότων και των παραβιάσεων, γιατί η Ουγγρική κυβέρνηση εξακολουθεί διαρκώς να μη σέβεται τους κανόνες, το δίκαιο και αυτό δεν έχει παρουσιαστεί ως φαινόμενο σε καμία άλλη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν καταρρύπτει το κράτος δικαίου και θα πρέπει κανείς να ζει στην Ουγγαρία για να καταλάβει τι συμβαίνει και ότι αυτό θα συνεχίσει όσο έχουν πλειοψηφία δύο τρίτων. Η κυρία Κούνα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο στόχος του άρθρου 7 γιατί φαίνεται ότι συνεχίζεται η καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ οι κυβερνήσει άλλων χωρών μένουν με τα χέρια σταυρωμένα και αδρανούν. Μέχρι πότε θα περιμένουμε. Πόσο θέλετε να σοβαρέψει η κατάσταση και να επιδεινωθεί για να κουνήσει το δαχτυλάκι της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να περιμένουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να κάνουμε αυτό που απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω που οφείλεται το πρόβλημα. Μήπως ε, οι κυβερνήσει των χωρών μελών φοβούνται ότι θα βρεθούν και αυτές στο στόχαστρο του ελέγχου κάποια στιγμή. Αν είναι αυτός ο φόβος του, τότε πραγματικά είναι υποκριτική η συμπεριφορά τους. Θα πρέπει να δράσουμε πάρα αυτά. Ιδεμή θα χάσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Στον επόμενο μιλητή θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο, επειδή βλέπω μία αυξημένη ε, διάθεση για μπλε κάρτες, όπως και αιτήματα για catch στην όντως σοβαρή συζήτηση, να πω ότι θα δέχομαι μία μπλε κάρτα για κάθε ομιλητή, αυτός που θα σηκώσει πρώτος την μπλε κάρτα. Και επίσης σημειώνω ότι ζητούν μπλε κάρτα συνάδελφοι που έχουν